Uh, Μάλιστα. Νομίζω ότι όσοι είναι να συμμετέχουμε στη συζήτηση που θα γίνει είμαστε εδώ. Έχουμε φτάσει στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, εξέταση των τροπολογιών. Σβέν, έχεις το λόγο. Okay, he's just booting up his uh, points. σαν σημειώσει του. I, I think uh, uh, we do it a bit differently. Λοιπόν, ας κινηθούμε λίγο διαφορετικά. Καταρχάς, με είναι ανοιχτό έτσι δεν είναι. Θα προσπαθήσω να μιλήσω γκλόμπις, μια κοινή σε όλους μας γλώσσα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις τροπολογίες σας πάντως. Δεν έχω ακόμα μπροστά τις σημειώσεις μου. Αυτό μπορώ να πω πάντως εν είδη εισαγωγή είναι ότι κινούμεθα όλοι πάνω κάτω στην ίδια κατεύθυνση. Θα ήθελα να χαιρετήσω τις διάφορες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί από τους συναδέλφους. Εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι διατηρούμε ένα παρόμοιο πνεύμα σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Όλοι ουσιαστικά θέλουμε να ενισχυθεί η αρτεκτονική εποπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς υπάρχουν σε κάποια σημεία κάποιες διαφορές, αλλά γενικά μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότερες απόψεις συγκλίνουν και αλληλοσυμπληρώνονται. Και αυτό αποκρισταλώνεται και στις τροπολογίες. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες σημαντικές διαφορές σε κάποια σημεία, αλλά ακόμα και όταν αυτές εντοπίζονται, δεν είναι οριζόντιες, αλλά αφορούν συγκεκριμένα σημεία και συγκεκριμένους ε, σκιώδεις συγητές που έχουν αποκλίνουσες απόψεις. Θα αναφερθώ σε κάποιες από αυτές. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε με την μακροοικονομική εποπτεία, Ενδεχομένως να έχετε δει ότι η αρχική μου πρόταση αναφέρεται σε ένα πλήρη διαχωρισμό μετά τη μελέτη που ζητήσαμε εμεί ως Επιτροπή και στη συνέχεια μετά τη μελέτη αυτή διέγραψα το δικό μου το αίτημα και ήρθα πιο κοντά στις δικές σας τις απόψεις που εξέφρασε το ΕΛΚ αλλά και άλλες πολιτικές ομάδες. Και έτσι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας. Υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι που λένε ότι οι δύο αυτές δομές θα πρέπει να είναι εντελώς ξεχωριστές, αλλά πιστεύω ότι πραγματικά μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση και να καταφέρουμε τελικά από κοινού να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία των δύο διαφορετικών αυτών δομών. Πάντως πρέπει ακόμα να κάνουμε μια περαιτέρω συζήτηση για το σημείο αυτό. Επίσης, είδα ότι υπάρχουν κάποιες σημαντικές διαφορές όσον αφορά το ζήτημα της δεσμευτικής διαμεσολάβησης. Ως προς αυτό, ορισμένοι συνάδελφοι θέλουν να ενισχύσουν τη δυνατότητα δεσμευτικής διαμεσολάβησης, άλλοι πάλι όπως ο Βόλφ θέλουν να περιορίσουν αυτή τη δυνατότητα. Ενδιαφέρουσες λοιπόν θα είναι και οι συζητήσεις και για το σημείο αυτό. Άλλοι πάλι όπως για παράδειγμα ορισμένοι από το ECR, θέλουν περισσότερες αρμοδιότητες διαμεσολάβησης για τις εποπτικές αρχές, αλλά δεν θέλουν να είναι διαμεσολάβηση αυτή δεσμευτική. Θέλουν να επισημοποιηθούν οι πιο άτυπες διαδικασίες, οι οποίες έχουν μια κάποια προστιθέμενη αξία και αυτό το είπαν και οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Από την άλλη όμως εγώ πιστεύω ότι υφίστανται ακόμα κάποια προβλήματα. Πρέπει η διαμεσολάβηση να είναι εν μέρη δεσμευτική και η δυνατότητα δεσμευτικής και μεσολάβησης είναι πολύ σημαντική προκειμένου να, έχουμε, να εγγυηθούμε, να διασφαλίσουμε και τις άτυπες αρμοδιότητες και εξουσίες. Τουλάχιστον η ε, τοποθέτηση αρχική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι, να είναι διαμεσολάβηση δεσμευτική για όλους τους τομείς, χωρίς να επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένα άρθρα του κανονισμού ή των οδηγιών. Επίσης να σας επενθυμίσω ότι ορισμένοι συνάδελφοι μας είχαν πει ότι έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ πολύπλοκο σύστημα και ότι ένα τέτοιο πολύπλοκο σύστημα τελικά δεν μπορεί να λειτουργήσει αρμονικά. Σε κάθε κανονισμό, σε κάθε οδηγία που εξετάζουμε, πολύ συχνά μιλάμε για το ζήτημα της δεσμευτικής διαμεσολάβησης και καταλαβαίνετε ότι μόνο και μόνο το ζήτημα αυτό από μόνο του κάνει γενικότερα την κοινοτική νομοθεσία αρκετά ακαμπτή. Έπειτα υπάρχει και το ζήτημα της παραβίασης της ενωσιακής νομοθεσίας Νομίζω πάντως ότι θα πρέπει να δώσουμε στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές τη δυνατότητα να επεμβαίνουν σε, όλη, όλο το φάσμα της κοινοτικής χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας. Και αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει είναι ότι αυτές οι εποπτικές, οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές δεν έχουν την υψηλή ισχύ και εξουσία που επιθυμούσαμε εμείς εξ αρχής να έχουν. Όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές, Πάλι νομίζω στα πλαίσια της Επιτροπής μας μόνο ο Βολφ Κλίντς θέλει να μειωθούν αυτές οι εξουσίες που απορρέουν από τις κατευθυντήριες γραμμές. Όλοι οι υπόλοιποι κινούμαστε στη διαφορετική κατεύθυνση. Και ξέρετε ότι υπάρχουν και ορισμένοι παράγοντες από τον ιδιωτικό τομέα που μας ζητούν να καταθέτουμε εμείς, να προτείνουμε κατευθύνες γραμμές μόνο να απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία για, την, για το χρηματοπιστωτικό τομέα. Ξέρετε όμως ότι ε, πολλές φορές εμείς ως νομοθέτες δεν είμαστε σε θέση να κινηθούμε με απόλυτη ευφυΐα, προορατικότητα και να δούμε τελικά πού θα εντοπιστούν τα προβλήματα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε κατευθυντήρες γραμμές οι οποίες δεν θα είναι δεσμευτικές μεν, αλλά για τις οποίες θα υπάρχει απαραίτητη αιτιολόγηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω εμεί να μην υποκύψουμε στην όλη πίεση που ασκείται αυτή τη στιγμή από τον ιδιωτικό τομέα, να πούμε ότι οι κατευθυντήριε γραμμέ αποτελούν μια μορφή ήπια νομοθεσία, soft law, και ότι θα πρέπει να διατηρηθούν. Λοιπόν, λυπάμαι, Βόλφ, αλλά δεν συμφωνώ για το σημείο αυτό μαζί σου. Τώρα, ως προς τις απόψεις της δικής μου πολιτικής ομάδας, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να περιοριστούν οι αρμοδιότητες του επόπτη αν εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι, αν δεν μπορούμε να επιλύσουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Πέρα από αυτά, προτείνονται κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες λύσεις από εσά κυρία Πρόεδρε, Ιδίω όσον αφορά κάποια διαδικαστικά ζητήματα, νομίζω ότι ε, σε ορισμένα σημεία πραγματικά πετούνται υψηλότατες γνώσεις νομομαθούς. Εγώ δεν θα μπορούσα μόνος μου να είχα καταλήξει τέτοιε προτάσεις. Συγχαρητήρια πραγματικά γιατί οι προτάσει που κάνετε είναι ιδιαίτερα ευφυεί και εξαιρετικέ από νομική ε, πλευρά. Φαντάζομαι ότι ε, θα έπρεπε να εντρυφήσετε πάρα πολύ στην κοινωτική νομοθεσία από νομικής πλευράς για να καταφέρετε να προτείνετε τόσο καλές προτάσεις. Ας σταματήσω πάντως στο σημείο αυτό. Ξέρω ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που εκκρεμούν και έχουν θίξει οι συνάδελφοι. Ξέρετε ότι έχουν υποβληθεί πολλές τροπολογίες, ε, οι οποίες σίγουρα θα μας επιτρέψουν να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις και συμβαστικές τροπολογίες για τα περισσότερα σημεία της πρότασης αυτής, προκειμένου να βοηθήσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει όντως να επεξεργάζεται την αναθεώρηση του ε, της πρότασης αυτής, προκειμένου πραγματικά να καταφέρουμε προς όλους τους παράγοντες του οικονομικού τομέα να δώσουμε τις απαραίτητες λύσεις. Σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας. Ευχαριστούμε οι σκιώδες εισηγητές τώρα με τη σειρά. Πρώτα λοιπόν εκ μέρους του ΕΛΚ η Άστριτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι καλή εδώ ευρωβουλευτής με την έννοια ότι συμμετέχω και παρακολουθώ Γι' αυτό λοιπόν όλο το Σαββατοκύριακο προσπάθησα να κοιτάξω τις 325 ε. τροπολογίες που υπέβαλαν οι συνάδελφοι μετά την παρουσίαση της έκθεσης του κύριου Γκίγκολτ. Και για να κερδίσουμε χρόνο θα σας πω ότι βρήκα λόγους που με ενθαρρύνουν, αλλά βρήκα και λόγους να μην είμαι τόσο αισιόδοξη. Θα ασχοληθούμε με την ουσία του θέματος αυτού τις επόμενες εβδομάδες και θα επανέλθουμε βέβαια. Όμως η έκθεση αυτή για το ευρωπαϊκό εποπτικό σύστημα δεν πρόκειται να καλύψει το κενό που υπάρχει ανάμεσα σε εμά, όπως παρατήρησε και ο εισηγητής, τα κενά κατανόησης δηλαδή ανάμεσα σε εμά και στο κοινό. Τώρα έρχομαι στη μεθοδολογία. Εδώ θα ήθελα να θυμώσω και θα εξηγήσω τι εννοώ. Από την πρώτη φορά που είχαμε ανταλλαγή απόψεων, είχα θέσει υπομφισβήτηση την χρησιμότητα του εγχειρήματο αυτού. Γιατί καλούμεθα να ψηφίσουμε ένα κείμενο που απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλη Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, ενώ θα έχει ήδη αυτή δημοσιεύσει αρχές Ιανουαρίου 2014 την έκθεσή της. Συνεπώς, οι συστάσεις μας θα ψηφιστούν εδώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει ήδη δημοσιεύσει τη δικιά της έκθεση. Οπότε, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει αφού δεν μπορούμε να τους επηρεάσουμε. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι στις τροπολογίες. Ομολογώ και εγώ ότι έχω πολλές αμφιβολίες εδώ για πολλούς λόγους. Διαπιστώνω πρώτα απ' όλα ότι ο εισηγητής είναι αυτός που έχει υποβάλει τις περισσότερες τροπολογίες. Έχει βέβαια κάθε δικαίωμα. Αλλά πρέπει να παραδεχτείτε ότι είναι λίγο παράδοξο να συντάσει κανείς μια έκθεση και μετά, μερικές εβδομάδες αργότερα, να υποβάλει ένα τόσο μεγάλο αριθμό τροπολογιών στο ίδιο αυτό θέμα που ο ίδιος ε, συνέταξε. Ο κύριος Γκικόλτ θα μου απαντήσει ότι ήθελε να λάβει υπόψη του τις ε, δικές μας ε, παρατηρήσεις και τους συσχετισμούς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εποπτεία. Οπότε θα σας πω ότι όταν παρουσιάστηκε η έκθεση αυτή, που σίγουρα θα κόστισε κάμποσα χρήματα στο Κοινοβούλιο, δεν ξέρω πόσα, ενώ παντού προσπαθούμε να κάνουμε οικονομίες. Όταν λοιπόν παρουσιάστηκε εδώ, ήμασταν πολύ λίγοι σε αυτή την αίθουσα, στην αίθουσα που συζητήθηκε. Κύριε Πρόεδρε, ο εισηγητής που έφτασε λίγο αργότερα και δύο σκιώδεις εισηγητές. Εγώ και πρόεδρος τους, τους σοσιαλιστές. Αυτό ήταν όλο. Και έφυγε και νωρίτερα ο εισηγητής. Συνεπώς, δεν είναι πολύ καλά όλα αυτά. Δεν δίνουν ωραία εικόνα. Φυσικά, μπορώ να αντιληφθώ τι θα απαντήσει ο εισηγητής, αλλά εκεί που πραγματικά δυσκολεύομαι, και αυτό δεν έχει να κάνει με τον εισηγητή μας αυτό καθ' αυτό, αλλά με όλους τους συναδέρφους, είναι ότι η έκθεση αυτή πρωτοβουλίας είναι υπερβολικά φορτωμένη με αιτιολογικές σκέψεις, με παρατηρήσεις που δεν είναι καν επαληθεύσιμες. Το αποτέλεσμα είναι να καταλήγουμε σε ένα εντελώς ε, δυσνόητο κείμενο όπου το δέντρο θα κρύβει το δάσος. Οι περισσότερες τροπολογίες τουλάχιστον που έχουν υποβληθεί αυτή την εικόνα παρουσιάζουν. Συχνά, κύριε Πρόεδρε, σε αυτήν την Επιτροπή προσπαθούμε να, είμαστε, να προσέχουμε τη λεπτομέρεια. Να φροντίσουμε οι νομοθέτες να μην επιβάλλουν μέτρα δεύτερου επίπεδου ή να μην επιβάλλουν, σε, να μην επιβάλλουν όργανα που δεν είναι τόσο δημοκρατικά, τις απόψεις τους ε, στα δημοκρατικά όργανα. Εν όμως το θέμα αυτό μπορούμε να το δούμε και ανάποδα. Η νομοθετική εξουσία πρέπει να παραμείνει νομοθετική. Και κατά τη γνώμη μου πρέπει να σεβόμαστε ό,τι λέει ο νόμος και έτσι οι νομοθετικές αρχές να ασχολούνται με τα νομοθετικά και οι ρυθμιστικές με τα ρυθμιστικά. Συνεπώς, μία κοινοβουλευτική έκθεση η οποία αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Εποπτικό Σύστημα για τις οικονομικές αγορές, πιστεύετε ότι πρέπει να αναφέρεται σε έλλειψη πραγματογνωμοσύνης για τα γεωργικά παράγωγα, για παράδειγμα. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που αναφέρονται σε τέτοιες λεπτομέρειες, σε τέτοια ειδικά ζητήματα, ακόμα και η δικιά σας δικές σας τροπολογίες αναφέρονται σε μικρές λεπτομέρειες που κατά τη γνώμη μου δεν έχουν δουλειά εδώ. Η δουλειά μας δεν είναι να κάνουμε άλλη μία έκθεση συμβουλευτικού χαρακτήρα. Εννοείται οι συγκητέ και ευρωβουλευτέ είναι ελεύθεροι να υποβάλουν ό,τι θέλουν ω τροπολογίε, αλλά με κάθε μετριοφροσύνη Θέλω να πω ότι έτσι δεν βοηθούμε ούτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε τη δικιά μας την Επιτροπή, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήγουμε σε μία έκθεση η οποία τελικά είναι ακατανόητη. Φυσικά κύριε Πρόεδρε η πλειοψηφία θα αποφασίσει εδώ. Πάντως, τις επόμενες εβδομάδες να ξέρετε ότι εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε η έκθεση αυτή να κρατήσει μια συνοχή και πολύ θα ήθελα οι συνάδελφοι που θα έχουν διαπραγματεύσεις μαζί μου να κατανοήσουν τη θέση μου και να τη συμμεριστούν κατά προτίμηση. Τη θέση μου και την ανησυχία μου που είναι να εκπονήσουμε μια σύντομη έκθεση, απαιτητική συγχρόνως, η οποία αναφέρεται σε αρχές και δεν χάνεται στις λεπτομέρειες. Ειλικρινά ελπίζω να εισακουστώ σε αυτό το σημείο. Επί της ουσίας, επιτρέψτε μου, να επανέλθω στην αρχή που έλεγα ότι δεν υπάρχει χάσμα μεταξύ μας που να μην μπορεί να καλυφθεί. Πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε από ό,τι ήδη υπάρχει. Και αυτά σιγά σιγά να τα τροποποιούμε. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Εποπτεία ήδη από μόνη της αποτελεί μια τεράστια αλλαγή. Συνεπώς, την αλλαγή αυτή να την παρακολουθήσουμε και να μην ακολουθήσουμε την αρχή, τα ξαναγράφουμε όλα από την αρχή. Όσον αφορά τώρα τις εποπτικές αρχές, εγώ πιστεύω ότι εδώ υπάρχει πλειοψηφία προκειμένου οι αρχές αυτές να γίνουν πιο ευρωπαϊκές και αυτό θα γίνει αν έχουν περισσότερες αρμοδιότητες management, αν ξαναδούμε τον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουν, ενώ η συγχώνευση πιστεύω ότι είναι μια πολύ πρόωρη ιδέα. Έρχομαι τώρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Και εδώ πρέπει να υπάρχει εξέλιξη κατά τη γνώμη μου. Δεν θα ήθελα όμως να χαλάσουμε αυτό που φτιάξαμε το 2010. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να υπερέχει στο όργανο αυτό, διότι κάνει καλά τη δουλειά της και διότι έχει την πραγματογνωμοσύνη που χρειάζεται. Κάτι το οποίο δεν είναι αυτοσχεδιασμός. Χτες άκουγα τον κύριο Ντράγκη που Κάποιοι τον ε, κατηγόρησαν ότι υπερβαίνει τα καθήκοντά της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι αλήθεια ότι η ΕΚΤ έχει όλο και πιο ενισχυμένες αρμοδιότητες. Ο πρόεδρος Δράγκη χτες απάντησε ότι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα πάντα όσον αφορά τη διαφάνεια για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. Δηλαδή συνειδητοποιεί ότι εδώ τίθεται θέμα της αξιοπιστίας της. Συνεπώς θα κάνει τα πάντα για να συμμορφωθεί στα όσα προβλέπονται. Και δεν έχω εγώ καμία αμφιβολία ότι όντως θα το κάνει. Στο μεταξύ είμαι κατά του να κοπεί η σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Θα σταματήσω εδώ. Ελπίζω να καταλήξουμε σε μια παρουσιάσιμη έκθεση, ευανάγνωστη και κατανοητή, η οποία να αντιστοιχεί στα όσα περιμένει ο κόσμος από ένα νομοθέτη και όχι μια εταιρεία ελέγχου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Λούλιν. Ο Αντολίν τώρα, εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Σας ευχαριστώ πολύ. 34 τοπολογίες κατέθεσα κάποιες από αυτές και με την Ελίζα Φερέρα από κοινού, συντονίστρια της ομάδας μας. Σημερίζομαι σε μεγάλο βαθμό το σχέδιο του Σβέν Γκίνγκολτ και που πιστεύω ότι συμπίπτω επίσης και με την αξιολόγηση σε μεγάλο βαθμό <clears throat> από το ίδιο το Κοινοβούλιο. Η δημιουργία Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας είναι μια διαδικασία ενρευστό που εξελίσσεται. Βρισκόμαστε σε μια πρώτη φάση. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή αυτή για να προβληματιστούμε και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Πιστεύω τρεις μεγάλοι προσανατολισμοί υπάρχουν. Ο πρώτος είναι η σχέση των ευρωπαϊκών αρχών εποπτείας με το ενιαίο σύστημα εποπτείας, ευρωπαϊκό σύστημα ε, εποπτείας. Και αυτό δεν αμφισβητεί θα έλεγα εγώ, δεν θέτει ένα αμφιβόλο τις αρχές εποπτείας τις ευρωπαϊκές, αλλά τις συμπληρώνει, τις ενισχύει για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αλλά έχει δημιουργήσει και κάποια, ας το πω έτσι, ε, μη συμβατότητα ή ασυνέχεια διότι σε σχέση με τις αρμοδιότητες ε, υπάρχουν εδώ πράγματα που διαφοροποιούνται σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας. Μελλοντικά θα πρέπει τη μέγιστη συνεκτικότητα να αναζητούμε σε σχέση με το αρχικό αυτό πρότυπο που θα εξελιχθεί προς το μέλλον. Υπάρχει και μια άλλη πτυχή που είναι ενδιαφέρουσα. Για πρώτη φορά υπάρχει το πρότυπο μακροεποπτείας σε σχέση με την μικροεποπτεία σε σχέση με το εγχείρημα μικροεποπτείας για την διασφάλιση ε, της ρευστότητας ε, ε, των τραπεζών και των ασφαλιστικών οργανισμών σε ένα πλαίσιο διάφανο όσον αφορά τις αγορές ε, αξιών και χρεογράφων αλλά για τη διαφάνεια νομίζω ότι πιστεύω ότι και για την υποστήριξη την επιμελητιακή και της γραμματείας τώρα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο αν η μακροεπιτήρηση, η μακροεποπτεία είναι απόλυτα συμβατή με την εντολή που είναι πολύ εξειδικευμένη για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα όσον αφορά την νομισματική σταθερότητα, τη σταθερότητα των τιμών. Να δούμε δηλαδή συγκεκριμένες πτυχές όσον αφορά το νομισματικό σύστημα προς την ανάπτυξη και την απασχόληση. Και έτσι πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε αν μπορεί εδώ να υπάρξει μια ε, παρέκκληση όσον αφορά αυτά τα θέματα από πλευρά της Ευρωπαϊκής. Πρέπει να το εντάξουμε περισσότερο μέσα στο σύστημα της οικονομικής ε, διακυβέρνησης ε, όπως γίνεται και στι ΗΠΑ σε σχέση με εμά, δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό έχω κάποιε προτάσει ώστε η μακροεποπτεία στι συστάσει μα, να ο έλεγχο με αυτέ τι συστάσει αφεαυτών να μπορέσουμε να διασυνδέσουμε αυτά τα θέματα με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την ανάπτυξη, την εξέλιξη της ε, ε, διακυβέρνησης στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια άλλη πτυχή είναι πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την λειτουργία των αρχών εποπτείας. Υπάρχουν κάποιες πτυχές λειτουργίας ή λειτουργικότητας εδώ που μπορεί να είναι θετικές. Ένα παράδειγμα. Οι αρμοδιότητες που θα μπορούν να δίνονται στην Προεδρία, θα έχει η Προεδρία αυτό νομίζω μπορεί να επιτρέψει μια καλύτερη λειτουργικότητα. Ένα χαρακτήρα πιο θα λέγαμε περισσότερο εκτελεστικού χαρακτήρα, πιο αποτελεσματική δράση, πιο άμεση, πιο ευέλικτη αν χρειαστεί σε διάφορες περιπτώσεις η συνολική ε, δράση να μπορεί να αναπτύσσεται συλλογικά αλλά και για την ανάπτυξη συγκεκριμένων στόχων να μπορεί η Προεδρία να δρά με ένα πλαίσιο ευρύτερης εντολής. Δεύτερο, νομίζω ότι είναι μια στιγμή όπου οι ενδιαφερόμενοι, οι stakeholders, οι εμπλεκόμενοι θα μπορούν να εκφραστούν για αυτή τη διαδικασία και να, να γίνεται αυτό με πιο ισορρόπο τρόπο και περισσότερο συλλογικά, να συμμετέχουν περισσότερο αλλά και να ενισχύσουμε τις επιτυχίες όσον αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία. Έχω υποβάλει προτάσεις σχετικά. Ένα άλλο θέμα είναι ποιες αρμοδιότητες και πώς μπορούν αυτές να αναπτυχθούν. Έχουμε το θέμα της ε, διαμεσολάβησης, της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης και ο σχεδιασμός για να επιλύονται αντιπαραθέσεις ή τριβές ώστε να μην είναι οι αρχές οι ίδιες ένας φορέας να μην είναι δικαστής και εμπλεκόμενος και δεν θα πρέπει λοιπόν να γίνεται οποιαδήποτε σύγχυση θα πρέπει να αναζητηθεί μια κοινοτική μέθοδος Νομίζω εξακολουθεί να ισχύει αυτό, αλλά η διαμεσολάβηση θα πρέπει να βρει μια συνάφεια και συνεκτικότητα σε σχέση και με την εποπτεία. Μπορούν σε πολλές περιπτώσεις όχι μόνο να έχουμε κάποιες τριβές αλλά μπορεί να υπάρχουν και διαφορές απόψεων που μπορεί να έχουν ε, ε, επιπτώσεις και γι' αυτό οι αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ανάληψης ιδίας πρωτοβουλίας να δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτό θα μπορεί να συνεισφέρει από πλευρά του για να διασφαλίζεται αυτή η συνεκτικότητα, η συνάφεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια άλλη πτυχή αναφέρεται στους καταναλωτές έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει ρητή κατηγορηματική εντολή γι' αυτό, αλλά θεωρούμε ότι καλό θα ήταν να κωδικοποιηθούν όλα αυτά που αφορούν την προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών. Είναι λοιπόν μια πτυχή αυτή που βρίσκεται εδώ και στοχεύει στις αρχές ε, να τύχει προσοχής και με την αναδιάρθρωση ή την δόμηση αυτή είναι η θετική στιγμή να κάνουμε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ένα τέτοιο προσανατολισμό να ακολουθήσουμε δύο νέες αρχές εισάγονται σε σχέση με τις αρχές εποπτείας της Βασιλείας τη συλλογική διακυβέρνηση και το θέμα της ε, διαφάνειας θεωρούμε ότι η ανάπτυξη αυτών των αρχών είναι πολύ σημαντική υπόθεση και πέρα από την συλλογική ολοκληρωμένη διαχείριση πρέπει να αποκτήσουμε και μια σημαντική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν θεσπίζουμε κανόνες για το bail-in στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανταποκρίνονται οι αρμόδιοι σε σχέση με τις ευθύνες που θα επομίζονται μέσα στο πλαίσιο της διακυβέρνησης. Το σύστημα διακυβέρνησης θα πρέπει να προσαρμοστεί και να αναδιαρθρωθεί μέσα στο πλαίσιο όλων αυτών των εξελίξεων. Και συνιστούμε λοιπόν αυτό να αποτελέσει τμήμα των ζητημάτων που πρέπει να τύχουν προσοχή από εμάς. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι η εποπτεία των υποδομών. Διασυνοριακά, cross-border υποδομές δηλαδή με άλλο, με άλλο τρόπο ε, διασυνοριακές, διαμεθοριακές. Πρέπει σαφώς να υπόκεινται άμεσα στην ευρωπαϊκή εποπτεία. Θεωρούμε είναι η πιο λογική μορφή και τρόπος για να αποφύγουμε να καταλήγουμε μετά σε, διε, σε επιδιατησία και να υπάρχουν ε, διαφορές και αποκλήσεις. Πρέπει να έχουμε κοινέ δόμες και αρχές για μια κοινοτική εποπτεία και προς αυτή την κατεύθυνση θα υποστηρίξουμε να κινηθούμε προς αυτό τον προσανατολισμό. Υπάρχουν και άλλα, αλλά αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Θέλω να επιμείνω και να εμείνω ότι οι προτάσεις αυτές που υποβάλλω είναι κίνητρα ώστε να βρούμε συμβιβαστικές διατυπώσεις με τον εισηγητή από τις έκθεσεις και να βρούμε δυνατότητα επίτευξης συνένεσης για το νομοθετικό μας έργο. Uh, Ευχαριστούμε. Ο Βόλφ, ευχαριστώ Σάρων. Ίσως να ξεκινήσω με αυτό το σημείο επί του οποίου άσκησε επικρίσεις ο Σβέν πιο πριν. Με το θέμα του αν οι εποπτικές αρχές υποχρεωτικά θα διαδραματίζουν ρόλο διαιτησίας, θα εμπλέκονται σε υποχρεωτική διαιτησία <clears throat> και θα υπονούν ε, δεσμευτικές ε, αρχές και κατευθύνσεις. Δεν είμαι καταρχήν εναντίον, αλλά από τον νομοθέτη στην πρώτη φάση θα πρέπει αντίστοιχα να ρυθμιστεί αυτό όπως το, βλέπουμε και τώρα το ότι ε, αυτά που αποφασίσαμε δεν θα το χαιρέτιζαν. γενικά δηλαδή ίσχυε κάτι τέτοιο αλλά εξειδικευμένα. Είδαμε στις αρχές του έτους ότι η ΕΣΜΑ και νομίζω ήταν σε συνάντηση με το χαρτοφυλάκιο Έμιρ ανέπτυξε, εξεπώνησε συστάσεις ή κατευθυντήριες γραμμές που τουλάχιστον προϋποθέτουν μια μερική τροποποίηση των όσων αποφασίστηκαν νομοθετικά στο πρώτο επίπεδο, level 1. Πρέπει να, να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Στο πρώτο επίπεδο, level 1, πρέπει να αποφασίζεται αν θα έχει δεσμευτική ε, ε, διατησία ή όχι ε, η αρχή αυτή. Τώρα όσον αφορά το ESRB έχω μια ολόκληρη σειρά παρατηρήσεων γι' αυτό. Πρώτον πρέπει να προσέξουμε το SRB, ε, το για την αντιμετώπιση συστημικού κινδύνου να μην επομιστεί ρόλους που δεν είχαν σχεδιαστεί γι' αυτό. Δηλαδή για το μακροπρόθεσμο, τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες σχεδιάστηκε και όχι για τις μικρότερες. Και γι' αυτό θα ήθελα να είμαστε επιφυλακτικοί να ε, υποβάλλονται σε σχέση με την υποβολή κάποιων προτάσεων να υπάρχει evaluation ή και άλλες δραστηριότητες. Ουσιαστικά είναι έργο ενός ε, εποπτικού τραπεζικού σώματος αυτά και δεν εντάσσονται, δεν εμπεριέχονται στο πεδίο ε, αρμοδιοτήτων ε, του SRB. Εγώ γι' αυτό θα ήθελα, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί στην νομοθετική διαδικασία, άμεσα να ενταχθεί. Μέχρι σήμερα, από ό,τι κατάλαβα, δεν, δεν είναι αυτή η εντολή που δίνεται Τίθεται το ερώτημα εδώ. Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε καταρτήσει, συγκροτήσει τα πράγματα για το SRB μετά από αρκετούς μήνες ε, εμπειρίας τώρα ανταποκρίνεται στην απόλυτη σοφία το, και είναι το τελεσίδικο στο οποίο καταλήγουμε. Είχαμε στο παρελθόν και για θετικούς λόγους θεωρήσει ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να είναι πρόεδρος εξίσου του SRB. Διαρωτώ με, αυτό σήμερα ανταποκρίνεται πραγματικά στην σοφία, στην απόλυτη σοφία ή μήπως ε, θα έπρεπε τα πράγματα να είναι πιο διαφορετικά. Ανεξάρτητα από το ε, ε, SRB θα παραμείνει εν όλο ή εν μέρη τμήμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τώρα να δούμε αν αυτό θα ενταθεί υπό τη στέγη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή όχι. Δεν είναι αυτό το αποφασιστικό για μένα. Το θέμα είναι να μην βρίσκεται τόσο άμεσα υπό την ίδια την επιρροή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ίσως. Και γι' αυτό όσον αφορά το άλλο θέμα συμφωνώ με τον εισήγητη ότι εδώ πραγματικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το μέγεθος των κρατών μελών. Τώρα, αν θα έχουμε μια απλή πλειοψηφία ή μια ενισχυμένη ε, πλειοψηφία που θα απαιτείται, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε για το Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορούμε να προβληματιστούμε γι' αυτό η πρόταση να είμαστε σε άμεση πιο ενδυναμωμένη επαφή με τους πολίτες αφενός είναι κάτι που μπορούμε να κατανοήσουμε και είναι κάτι επενέσιμο ως πρωτοβουλία αλλά δεν είναι λειτουργικό αυτό να έχει κάθε πολίτης άμεσα τη δυνατότητα να στρέφεται στην εποπτική αρχή που θα καταλήξουμε αυτή η δυνατότητα δηλαδή θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερβολικό φόρτο εργασίας και θα μπορούσε μόνο τότε να αντιμετωπιστεί από την εποπτική αρχή αν βρισκόταν ένα σύστημα λειτουργικό frequently asked questions and answers συχνά διατυπούμενες ερωτήσεις και απαντήσεις ώστε να μπορούν, ας το πω έτσι, να ε, επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα οι παρεμβάσεις και όχι επί παντός του επίστητου. Συμφωνώ απόλυτα και είναι σημαντικό αυτό, συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η εποπτική αρχή θα πρέπει να είναι αποφασιστική σημασία ε, να έχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται. Στο παρελθόν ήταν πρόβλημα αυτό. Η ανταλλαγή διασυνοριακά των πληροφοριών και της ενημέρωσης δεν λειτουργούσε καλά. Και εδώ έχουμε πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ταυτόχρονα πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε και ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας όλων αυτών για να αποφύγουμε ότι η επιβάρυνση που θα απορρέει από πλευράς εργασίας από όλα αυτά τα θέματα, συλλογή στοιχείων, ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και θεσμών, θεσμικών οργάνων, να μην οδηγεί σε δημιουργία γραφειοκρατικού βάρους και εμποδίων. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, πρέπει να τα εξετάσουμε πολύ καλά για να πάνε τα πράγματα σωστά. Διερωτώ με πέρα από αυτά πως οι εποπτικές αρχές μπορούν να έχουν την ανεξαρτησία που πρέπει να έχουν και να, απολαμβάνουν αυτής. Συνδέονται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε πολύ στενή επαφή με τις εθνικές εποπτικές αρχές που και μέλη αυτών ε, βρίσκονται σε αυτό το θεσμικό όργανο και ακούσαμε ότι οι εκπρόσωποι των εθνικών θεσμικών εποπτικών οργάνων σε σχέση με την ΕΣΜΑ για α το πω έτσι πολύ μικρό περιθώριο ελιγμών και κινήσεων αφήνουν και αυτό ουσιαστικά θα έπρεπε να το ξαναδούμε. Εδώ το ερώτημα λοιπόν το ζήτημα ποιο είναι. Η ανεξαρτησία διασφαλίζεται λοιπόν με αυτόν τον τρόπο όπως θα έπρεπε ή όχι. Η ανεξαρτησία φυσικά συνδέεται και με κάτι άλλο. Αν οι πόροι, τα κονδύλια είναι επαρκή ή όχι. Και συμφωνούμε ότι ακόμα οι πόροι, τα κονδύλια δεν επαρκούν ακόμα. Και όλη η δυνατότητα στελέχωσης από πλευρά στελεχών μιας ε, ενός θεσμικού οργάνου διαδραματίζει μόνο θεωρητικά ένα ρόλο, διότι αν δεν υπάρχουν και όταν δεν υπάρχουν τα κονδύλια δεν μπορεί κανείς να είναι ανεξάρτητος και να λειτουργήσει μέσα σε ένα αυτοτελές ε, ανεξάρτητο πλαίσιο. Αυτές είναι οι κυριότερες παρατηρήσεις μου. Έχω ένα και ίσονο σημασία εδώ που κάπου το έθιξες εσύ Σβέν πιο πριν. Το θέμα δηλαδή αν η παραβίαση κοινοτικού δικαίου πραγματικά επαρκώς εξετάστηκε σε αρκετό βάθος ή όχι. Προτού τώρα εγώ καταλήξω στο συμπέρασμα και πω ότι οι ανακριτικές ή διακριβωτικές δυνατότητες ε, των εποπτικών αρχών είναι περιορισμένες, θα ήθελα πριν πω κάτι τέτοιο να εξετάσουμε και να δούμε αν οι δυνατότητες που υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή πλήρως εξαντλούνται και χρησιμοποιούνται. Γιατί αν όχι τότε μπορούμε να δούμε τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια παραπέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εκ μέρου των Ευρωπαίων Συντηρητικών. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχει συνένεση μεταξύ πολλών σκιωδών. Είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο, οπότε συμφωνώ με την κυρία Λούλινγκ ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε την αρχική νομοθεσία όσον αφορά την ευρωπαϊκή εποπτεία. Οι τρεις αρχές ε, μεταρρυθμίζονται πολύ γρήγορα μετά την αρχή της εντολής τους. Η συγχώνευση πρέπει να οδηγήσει σε μια επιτυχή αρχή. Συμφωνώ πάντως ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα, ότι ήδη έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν οι προδιαγραφές εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε σίγουρα χρειάζεται και ο συντονισμός μεταξύ των 28 πλευρών. Υπό το φως αυτό λοιπόν έρχονται και οι τροπολογίες μου. Αρχίζω με την ανεξαρτησία της αρχής. Δεν πρέπει να αποδυναμωθεί ο ρόλος των ε, αρχών όσον αφορά το συντονισμό, βάζοντάς τες να ασχολούνται με καθημερινά θέματα, γιατί έτσι θα μπορούν λιγότερο να έχουν μια συνολική εικόνα των αγορών. Τώρα για τον προϋπολογισμό και την μόχλευση. Πάλι εδώ το απορρίπτουμε γιατί φοβούμαστε ότι αυτό θα πλήξει την ανεξαρτησία. Οι τροπολογίες μου πάντως πάνε προς τη γραμμή που λέει ότι περισσότεροι ειδικοί να βοηθήσουν, ναι, αλλά πάντα να έχουμε υπόψη μας την ενίσχυση της ανεξαρτησίας. Ό,τι συμβουλές δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι συμβουλές αυτές και η διαφοροποίησή τους, δηλαδή κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλείνει από τις συμβουλές πρέπει να οδηγήσει και σε κάποια αιτιολόγηση. Να εξηγούν γιατί το κάνουν αυτό. Υπάρχουν και άλλα θέματα ανεξαρτησίας, τα οποία αναφερθήκαμε για το κατά πόσο κάνουμε την διάκριση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τον Πρόεδρο της Αρχής. Όλα αυτά είναι ευαίσθητα ζητήματα. Μην ξεχνάμε ότι έπρεπε να τροποποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Οπότε και εδώ πρέπει να προσέξουμε πολύ τις εποπτικές αρχές και να λάβουμε υπόψη μας τις χώρες που είναι μέσα και έξω από την Ευρωζώνη. Κάτι άλλο που θέλω να τονίσω, πέρα από την ε, ανεξαρτησία, πρέπει να δούμε τι γίνεται με την έρευνα παραβιάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας. Εμείς θα θέλαμε να ενισχυθεί αυτό και άλλοι εδώ το ίδιο. Οι εξουσίες που ήδη υπάρχουν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα. Πάντως συμφωνώ ότι Εκεί που οι ευρωπαϊκές αρχές πρέπει να επικεντρωθούν επίσης περισσότερο είναι στους καταναλωτές, είτε πρόκειται για πελάτες τραπεζών, είτε για οτιδήποτε άλλο πρέπει να επικεντρωθούν οι αρχές αυτές περισσότερο στους καταναλωτές ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι είναι σε πολύ καλή θέση οι ευρωπαϊκές αυτές αρχές για να το κάνουν. Πολλέ τροπολογίε μπορούμε να τις υποστηρίξουμε, γιατί προσπαθούν να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Αρχών και την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, προκειμένου να ενισχυθεί ακριβώ ο ανταγωνισμός. Και να μην υπάρχουν πια πρακτικές που να μην είναι θεμητές με τον ανταγωνισμό. Γιατί αυτό είναι σε βάρος των καταναλωτών. Γι' αυτό λέω ότι εδώ οι ευρωπαϊκές αυτές αρχές μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Και αλλού όμως θα θέλαμε να γίνουν πράγματα που θα βοηθήσουν περισσότερο τις ευρωπαϊκές αρχές στο έργο τους. γνωμοσύνη Πιο ενεργός ρόλος στις εκθέσεις αντικτύπου. Μελέτη κόστους-οφέλους για να έχουμε τα σωστά αριθμιστικά πλαίσια. Και να μπορέσουμε έτσι εμείς ως νομοθέτες να έχουμε τα στοιχεία που μας χρειάζονται για να βελτιώσουμε τα νομοθετικά μας κείμενα. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας προσφέρει τέτοια οικονομική ανάλυση με ανεξάρτητο τρόπο, είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε όλοι, γιατί θέλουμε οι οικονομικές μας νομοθετικές πράξεις να βασίζονται ακριβώς σε στοιχεία, σε αποδείξεις. Στηρίζω πάντως όλα τα μέτρα που θέλουν να ενισχυθεί η διαφάνεια. Κυρίως ο τρόπος με τον οποίο οι ευρωπαϊκές αρχές ε, συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή με τα άλλα θεσμικά όργανα. Εν κατακλείδη πιστεύω ότι είναι σωστή κίνηση που κάνουμε, ότι λειτουργούν καλά. Οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν φτιαχτεί για τον σωστό σκοπό, οπότε δεν θα ήθελα πλήρως να αλλάξουν. Να διασφαλίσουμε όμως ότι χρησιμοποιούν όλες τις αρμοδιότητες που έχουν αποτελεσματικά, κυρίως όσον αφορά την έρευνα και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Θέλω να ενισχυθεί παρετέρω η ανεξαρτησία τους, να μην μειωθεί αυτή λόγω παρεμβάσεων του κλάδου και θέλω επίσης να επικεντρωθούν περισσότερο στην προστασία των καταναλωτών, υποστηρίζουν τους καταναλωτές πιο πολύ, ε, περισσότερο και λιγότερο τους παρόχους υπηρεσιών. Κατά τα άλλα, είναι πολύ νωρίς, μέχρι τώρα πάντως τα έχουν πάει καλά και θα ήθελα οι αρχές αυτές να χρησιμοποιήσουν τις αρμοδιότητες που εμείς πιστεύουμε ότι τους έχουμε δώσει πριν τις αναδιαρθρώσουμε πλήρως και τις μεταρρυθμίσουν. Κάνουν καλή δουλειά και πρέπει να τις στηρίζουμε. Η συγχώνευση είναι πρώιμη. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Και εγώ είμαι στον κατάλογο μιλητών. Υπάρχει κανένα άλλος που θέλει το λόγο? Όχι. Να συνεχίσω. Σε ευχαριστώ Σβέν για το σχέδιο έκθεσης και θα ήθελα να δω και όλες τις υπόλοιπες ε, τροπολογίες. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να τις διαβάσω όλες ακόμα. Τώρα οι δικές μου τροπολογίες είχαν ως στόχο να ενισχύσουν ανεξαρτησία των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών και τον τρόπο που λειτουργούν σε καθημερινό επίπεδο και αναφέρθηκα επίσης και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το διορισμό των επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και θυμάστε ότι αρχικά είχαμε αντιμετωπίσει εκεί κάποια προβλήματα. Και επίσης ε, υποστηρίζω και όλη την ρυθμιστική ατζέντα που προβλέπετε για τις αρχές αυτές. Λυπάμαι Σβέν αν ε, χρειάστηκε να αναλύσεις όλα αυτά τα πολύ ε, διαδικαστικά ζητήματα, τα οποία ενδεχομένω να φανίζονται κάπως ε, φορτικά, αλλά χρειάστηκε εγώ να επισέλθω στα ζητήματα αυτά. Στις τροπολογίες 8 και 84 θέλω να εξασφαλίσω ότι οι διαδικασίες των εποπτικών συμβουλίων δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τα συμφέροντα των κρατών μελών από πλευρά συμβουλίου αντιμετωπίζουν πολύ συχνά τα εποπτικά συμβούλια ως μίνι συμβούλια και πολλές φορές εκπροσωπούν εκεί πέρα κράτη-μέλη. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι τα εποπτικά συμβούλια να ακολουθούν λίγο πιο πολύ την κοινοτική μέθοδο, το ευρωπαϊκό σύστημα οι ε, συμμετέχοντες δεν θα πρέπει να εκπροσωπούν στα συμβούλια αυτά εθνικά συμφέροντα γιατί υπονομεύεται και η ανεξαρτησία και η αξιοπιστία του όλου υποπτικού συστήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ένα, μια ευρωπαϊκή διάσταση στα συμβούλια αυτά καθότι πολλές φορές ξέρετε ότι συμμετέχουν σε διεθνείς διαπραγματεύσεις και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση σε διάφορες επιτροπές διεθνείς όπως η Επιτροπή της Βασιλείας. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να μιλάμε πιο στεναρά, εκφράζοντας όμως τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Αυτό δεν το είχαμε εξασφαλίσει από την αρχή και χρειάστηκε να κάνουμε κάποιες διορθώσεις, όπως για παράδειγμα στις διαπραγματεύσεις που γίνανε για τις οδηγίες για, την, για τα κεφάλαια τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι τράπεζες. Επίσης, όσον αφορά το διορισμό των προέδρων των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, θέλω να αποφύγουμε οποιαδήποτε διάκριση μπορεί να υπάρχει. Είδαμε ότι είχε γίνει κάτι τέτοιο σε σχέση με την ηλικία στο παρελθόν. Προφανώς δεν θέλουμε να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Έχω υποβάλει κάποιες σχετικέ τροπολογίε. επίσης τροπολογίε όσον αφορά την κοινή επιτροπή. Θέλουμε να αποφύγουμε εδώ πέρα οποιαδήποτε επικάλυψη εργασίας και καλύτερο συντονισμό μάλιστα τη εργασία. Και κάποιες τροπολογίες έχουν να κάνουν και με την εξαρτησία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω είπε και η ΚΕΙ, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη προφανώς τη γνωμοδότηση των Ευρωπαϊκών Υποπτικών Αρχών, αλλά να μπορούμε και εμείς μετά ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ελέγχουμε την όλη κατάσταση. Προφανώ εξελίσσονται συνεχώ οι διαδικασίε αυτέ και θα έλεγα ότι σε πολλέ περιπτώσει βελτιώνονται μάλιστα. Έχω αποβάλει και κάποιε τροπολογίε στι οποίε ε, λέω ότι θα μπορούσαν οι ευρωπαϊκές υποπτικές αρχές να καταρτήσουν κάποιες δείκτες επιδόσεων όσον αφορά την καθημερινή εποπτεία που κάνουν και θα μπορούσαν επίσης να κάνουν και κάποιες οικονομικές αναλύσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ενδεχομένως βέβαια για να κάνουν κάτι τέτοιο θα χρειαστούν και επιπλέον πόρους. Ωστόσο πρέπει να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε και αυτές τις επιβλέψεις όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Οι ευρωπαϊκές οπτικές αρχές μπορούν να επιτελέσουν και εκεί έναν επικοδομητικό ρόλο είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τον ρόλο και την προάσπιση των καταναλωτών ως προς τις αγορές. Προφανώς οι ευρωπαϊκές οπτικές αρχές μπορούν να έχουν κάποιο ρόλο, αλλά αυτό που βλέπουμε πολλές φορές είναι ότι οι ρυθμιστικές αρχές των αγορών λαμβάνουν το ρόλο αυτό. Γι' αυτό τον λόγο θέλουμε να ενισχύσουμε τις ε, κυρώσεις που θα πρέπει να επιβάλλονται για παράδειγμα στα πλαίσια της MIFID σε σχέση με την CRD4. Ξέρετε, όταν διαπραγματευόμασταν τη CRD4, το Συμβούλιο ήθελε να μειώσει τις κυρώσεις του προληπτικού ελέγχου. Όσον αφορά τώρα τις έδρες των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αυτών Αρχών, πολλοί έχουν αναφερθεί στο ζήτημα αυτό, εγώ όμως όχι. Θεωρώ ότι προσπαθείτε μέσω τροπολογιών αυτών να αποστείλετε ένα πολιτικό μήνυμα. Δίστανται οι απόψεις, πολλές φορές οι απόψεις έχουν προσωπικό χαρακτήρα. Δεν μπορούμε όμως να λέμε ότι εξαιτία της έδρας δεν συνεργάστηκαν καλά οι Ευρωπαϊκές Οπτικές Αρχές. Το αντίθετο θα έλεγα εγώ. Είχαν καλή συνεργασία οι αρχές αυτές μεταξύ τους. για μένα είναι σαφές ότι λειτουργούν από κοινού. Όπως και άλλοι συνάδελφοι, έτσι και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αναλύσουμε ακόμα περισσότερο το ρόλο που θα πρέπει να έχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Σίγουρα επικρατεί πάρα πολύ στα πλαίσια του Συμβουλίου αυτού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Σαφώς θα μπορούσε το Συμβούλιο αυτό να ακούει και τα όσα έχουν να πούν οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό αυτό Συμβούλιο κάτι διαφορετικό. Να μπορέσουμε δηλαδή να έχουμε μια πιο ευρεία προσέγγιση της αντιμετώπισης του συστημικού κινδύνου. Οι κεντρικές τράπεζες σκέφτονται και λειτουργούν σαν κεντρικές τράπεζες στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης δεν καταφέραμε να αποφύγουμε τον πολύ ε, αρνητικό ρόλο που ε, είχαν οι συνήθεις ύποπτοι στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να έχουμε ένα συμβούλιο το οποίο θα έχει μικρότερη διάσταση, θα έχει ένα μικρότερο σχήμα, θα μπορεί να συνεδριάζει πολύ πιο συχνά και θα μπορεί να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις. Και θεωρώ βέβαια ότι με τους, τους ισχύοντες περιορισμούς, το Συμβούλιο αυτό και παρά τις αντικσότητες που αντιμετώπισε λειτουργεί σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει όμως την απαραίτητη αυτή δομή που θα το επιτρέψει να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και προς αυτό θα πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό, θα προχωρήσουμε σε λίγο σε ψηφοφορίες και δίνω τώρα πάλι το λόγο στον εισηγητή, στον Σβέν. Ευχαριστώ. Για να απαντήσω σε κάποιες παρατηρήσεις. Με τις τροπολογίες σας, Πρόεδρε, συμφωνώ γενικά μιλώντας. Συμφωνώ ότι υπάρχουν κάποια θέματα πάνω στα οποία τελικά θα διαφωνήσουμε. Είναι το θέμα της έδρας, το θέμα του κατά πόσο πρέπει να είναι σε, μία, σε ένα μέρος, σε μία τοποθεσία όλες αυτές οι αρχές ή όχι και τελικά μπορεί να μην συμφωνήσουμε και την ψηφοφορία των κανόνων. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τεθούν σε ψηφοφορία με τους κανόνες που ισχύουν εδώ. Το ότι υπάρχουν διαφορές υπάρχουν. Τι να κάνουμε. Πάντως δεν συμφωνώ ότι η δημοκρατική ψηφοφορία έχει να κάνει με το μέγεθος των αγορών. Η ψηφοφορία έχει να κάνει με τους ανθρώπους, δεν έχει να κάνει με τα ευρώ ή με το νόμισμα το οποίο έχετε. Πάντως, ό,τι συζήτηση και να κάνουμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε το ευρύτερο θέμα. Συμφωνώ με την ΚΕΙ και με την Πρόεδρο για το ότι η προστασία των καταναλωτών πρέπει να ενισχυθεί. Αυτό έχει να κάνει και με τις τράπεζες και με τις ασφάλειες και νομίζω ότι υπάρχουν προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο οι αρχές αυτές δρούν. Βέβαια, όταν αρχίσει να ισχύει η MIFID, τότε θα έχουν επιπλέον αρμοδιότητες για την προστασία των καταναλωτών. Το βασικό θέμα το έθεσε η Άστριτ. Σε τι βαθμό πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες και μήπως δημιουργείται σύγχυση εξαιτία του μεγάλου αριθμού τροπολογιών που κατέθεσε αυτός ο κακός εισηγητής. Συγγνώμη Άστριτ, οι τροπολογίες αυτές έρχονται και από τις τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Δεν είναι μόνο από μας. Και εκείνοι μας ζήτησαν να υποβάλουμε τέτοιες τροπολογίες. Προσπαθώ να λάβω υπόψη μου στα σοβαρά τις δικές τους παρατηρήσεις. Πάντως συμφωνώ ότι οι τροπολογίες πρέπει να οδηγήσουν σε ένα κείμενο που να διέπεται από συνοχή και να είναι κατανοητό και γι' αυτό μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε. Θα προσπαθήσω προς αυτή την κατεύθυνση να εκπονήσω συμβαστικές τροπολογίες. Αλλά δεν έχει νόημα να κάνουμε μελέτες, να ζητάμε μελέτες τις οποίες μετά δεν χρησιμοποιούμε για να εκπονήσουμε την νομοθεσία μας. Και δεν φτάνει να μένουμε στο επίπεδο των αρχών, γιατί αυτό μπορεί να είναι καλό όταν αρχίζεις νέα νομοθεσία. Τώρα όμως χρησιμοποιούμε την εμπειρία που έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα. Και αν θέλουμε να μας πάρουν στα σοβαρά πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και λεπτομερείς. Βέβαια καλά διαρθρωμένο πρέπει να είναι το κείμενο και κατανοητό. Αυτά. Ελπίζω το στόχο αυτό να τον πετύχουμε όλοι μαζί, Πρόεδρε. Έπειτα. Υπάρχει και το θέμα που έθεσες εσύ, Κέι, για την σημασία που έχει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Και βλέπω στις τροπολογίες σου και κάποια ένταση. Εγώ λέω ναι, να μπορούν ο πρόεδρος να ξεκινάει κάποιες ερευνητικέ διαδικασίες, συλλογή δεδομένων ή κάτι άλλο, για να εξετάζεται η παραβίαση ακριβώς της κοινοτικής νομοθεσίας. Αν θυμάμαι καλά τη δικιά σου τροπολογία, εσύ θέλεις αυτές τις επιπλέον εξουσίες να τις περιορίσεις αυτές τις αρμοδιότητες του Προέδρου. Και εδώ βλέπω αντίφαση γιατί το πρόβλημα με τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές είναι ότι οι αρχές αυτές έχουν αρμοδιότητες μεταξύ άλλων και την εξέταση παραβιάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας, αλλά να χρησιμοποιήσουν τις αρμοδιότητες τους αυτές, χρειάζεται το Συμβούλιο Εποπτικών Αρχών να συμφωνήσει. Και άρα χρειάζεται να μείνει Συμβούλιο που θα συμφωνήσει. Αλλά εκεί συνήθως δεν συμφωνούν μεταξύ τους αυτό έχουν δείξει οι μελέτες μας. Και από αυτού προσπαθώ να βρω μια λύση. Πώς δηλαδή οι αρμοδιότητες αυτές θα τίθενται σε εφαρμογή χωρίς να πρέπει να προηγηθεί αυτό το μήνυ συμβούλιο. Αυτό πρέπει να εξετάσουμε και να λύσουμε. Αλλιώς θα έχουμε στη διάθεσή μας ευρωπαϊκές αρχές που θα έχουν αρμοδιότητες τις οποίε όμω δεν θα χρησιμοποιούν ποτέ. έτσι στις παραβιάσεις κοινοτικής νομοθεσίας δεν θα μπορούν να, κάνουν τίποτα. Το ίδιο ισχύει και με την δεσμευτική διαμεσολάβηση. Ακόμα κι αν υπάρχουν τέτοια θέματα στην νομοθεσία, πρέπει προηγουμένως να υπάρξει μια συμφωνία για να ξεκινήσει η διαδικασία. Αυτό εμποδίζει τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και μην το ξεχνάμε. Συμφωνώ με τον Αντολίν ότι χρειάζονται περισσότερες μακροοικονομικές ε, εξουσίες. Ο Σκίνερ, πώς το είπα, θα ζήτησε παραπάνω εξουσίες. Συμφωνώ για την ε, Μικτή Επιτροπή, Πρόεδρε. Τα είπε πολύ καλά η συμπατριώτησά σας, κύριε Σκίνερ. Υπάρχουν 8 δυνατότητες για βέτο προκειμένου να ληφθεί απόφαση. Υπάρχει και το θέμα της ενημέρωσης και των πληροφοριών. Βολφ, νομίζω ότι εδώ πρέπει να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει, γιατί από τη μια έχουμε το πρόβλημα ότι συχνά οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές δεν έχουν την αρμοδιότητα να ενημερωθούν. Πρέπει να ρωτούν το Συμβούλιο και από την άλλη οι αρχές αυτές υποβάλλουν ερωτήσεις. Οι εθνικές αρχές επίσης και στο μέλλον μπορεί να υπάρξουν και παραπάνω σώματα και τελικά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χρειάζονται πάρα πολύ προσωπικό απλώς και μόνο για να δίνουν τις πληροφορίες που τους ζητάνε οι διάφορες αρχές. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Όσον αφορά τώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Αυτό που μα έλεγε χθε ο Μάριο Τράγκε το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί λίγο πολύ είπε ότι υπάρχει πρόβλημα με το ότι έχουμε πολλά στο ίδιο σημείο. Το κατά πόσο πρέπει να διαχωριστούν ή όχι, πρέπει να το δούμε. Ακόμα και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ακόμα και αν όλοι συμφωνούμε ότι αποτελεί το θεσμικό όργανο κλειδί το οποίο μας βοήθησε να κρατήσουμε το ευρώ, συγχρόνως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι 24 ώρες το 24 ώρο μπορεί να δουλέψει ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όχι παραπάνω. Σε αυτή την κρίση προφανώς δεν μπόρεσε να δουλέψει όπως θα έπρεπε αυτό μπορεί να είναι μια απάντηση στην υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων. Θα σταθώ εδώ. Έτσι κι δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα, αλλά έχουμε την ψηφοφορία στην ημερήσια διάταξη, γι' αυτό σταματάω. Ευχαριστώ, Σβέν. Προσβλέπουμε στο να δούμε το τι θα γίνει με τις συμβαστικές τροπολογίες μεταξύ μας. Καταφέραμε πάρα πολλές ε, διαφορετικές ιδέες ε, να παρουσιάσουμε, να διατυπώσουμε και εξετάζονται και από την Επιτροπή συνολικά όλα αυτά. Πρέπει να προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο σημείο. Α, όχι, πρέπει να σας πω ότι θα ψηφίσουμε στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή στις 23 Ιανουαρίου, στοχεύοντας να περάσει στην περίοδο συνόδου του Φεβρουαρίου στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο το θέμα αυτό. Περνάμε τώρα European Investment Bank. Εντάξει. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι το σημείο 10. Εξέταση τροπολογιών για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εισηγητής ο κύριος Μπέρμαν. Δεν παρίσταται όμως. Υποθέτω ότι δεν είναι επίμαχο το θέμα μεταξύ μας αυτό σχεδόν εισηγητών του Τάις Μπέρμαν και πρέπει όμως να εξεταστούν αυτά τα θέματα θα περάσουμε στην ψήφιση άμεσα στη συνέχεια. Κάποιος θέλει να παρέμβει για τις τροπολογίες για αυτό το θέμα. Υποθέτω ότι η σιωπή είναι όχι, είναι άρνηση. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια παρέμβαση. Εσείς θέλετε να παρέμβετε, Βέρνα, Βέρνα Λάγεν. Ναι, νομίζω ότι πραγματικά δεν είναι επίμαχο αυτό το θέμα αυτής της έκθεσης του συναδέλφου. Τώρα θα ψηφίσουμε αμέσως στη συνέχεια. Ο κατάλογος, ο πίνακα ψηφοφοριών έχει συμφωνηθεί σε μεγάλο βαθμό μεταξύ μας. Η γνωμοδότηση νομίζω συνολικά είναι ισορροπημένη και η επικέντρωση στην αηφόρο ανάπτυξη είναι δεδομένη και είναι μεταξύ όλων των σημαντικών αυτών ετοιμάτων που διατυπώνουμε έχουμε τις τροπολογίες αυτές που ε, συμπεριλαμβάνουν αυτά τα αιτήματα και μπορούμε έτσι να ψηφίσουμε προς έγκριση. Επικέντρωση σε πράσινα σχέδια και προγράμματα όπως ε, ζητείτε από κάποιες ε, τροπολογίες το απορρίπτει αυτό η δική μας ομάδα. Ευχαριστώ. Okay, θέλει να παρέμβει παρακαλώ. Κανείς. Ε, τότε πολύ ωραία. Αυτό σημαίνει ότι είναι σχετικά συνενετικό το θέμα αυτό. Τώρα, στη συνέχεια θα πρέπει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα γίνεται ώστε να υπάρχει και ο μεγαλύτερος αριθμός συναδέφων εδώ σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα για το 2014 για τις συνεδριάσεις της ΕΚΟΝ που υιοθετήθηκε το Σεπτέμβριο από πλευράς μας υπενθυμίζεται ότι λόγω των ναι, δεν θέλω πραγματικά. Πριν από τις ε, ψηφοφορίες θα το κάνουμε, ώστε να ακούσετε, να παρακολουθήσετε τις ε, ανακοινώσεις Προέδρου. Και σε σχέση και τώρα με τα όσα απαιτούνται από τις ε, διατάξεις, υπενθυμίστε ότι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα αρχικά είχαμε προβλέψει για τις 20 και 21 Ιανουαρίου μια εκδήλωση. Θα γίνει την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου τώρα αυτή η συνάντηση από τις 3 έως τις 6.30. Διακόπτεται η Πρόεδρος. Right, Λοιπόν θα συνεχίσω εντάξει. Όταν υπάρξει ησυχία Επίσης και στις 23 Φεβρουαρίου από τις 9 στις 12.30 και μετά από τις 3 έως 6.30 το απόγευμα και συνεδριάσεις τη κοινοβουλευτική επιτροπή θα επικαιροποιηθούν ε, στην ιστοσελίδα τα στοιχεία για αυτέ τις συνεδριάσεις. Σε σχέση και με πολιτική συμφωνία υπό την προϋπόθεση τεχνικής ε, ε, συμφωνίας επί των τεχνικών θεμάτων όπως καταλήξαμε, η οδηγία, η οδηγία θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2015 και θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2016 το σύστημα αυτό να λειτουργεί. Μια τελική συνεδρίαση και χθες και σήμερα υπό εξέλιξη διακόπτη πρόεδρος. Σταματώ συνέχεια όταν γίνεται, δημιουργείται φασαρία, θόρυβος και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Θέλετε λοιπόν να προχωρήσουμε, να ψηφίσουμε, σταματήστε τις συζητήσεις για να ολοκληρώσουμε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, εντάξει. Μια τελική τεχνικού χαρακτήρα συνεδρίαση βρίσκεται υπό εξέλιξη. Η επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 70 θα γίνει όταν θα έχει ετοιμαστεί το κείμενο αυτό και δεδομένη της ψήφιση στην Ολομέλεια προβλέπεται το Φεβρουάριο στην περίοδο συνόδου. Θα μπορούσε και να υπάρξει και κάποια αλλαγή για την κοινή ψήφιση κειμένων και σε σχέση με την, ε, ε, το τι θα ισχύσει ίσως υστερότερα σήμερα θα το γνωρίζουμε όμως ε, σε σχέση με την δεύτερη ανάγνωση θα μπορούσε να επιτευχθεί το Φεβρουάριο για τους τριμερείς διαλόγους MIFID ένας ενδέκατος διάλογος έγινε στις 12 Δεκεμβρίου για τις, τα παράγωγα και όσον αφορά το καθεστώς τρίτων χωρών πρόσβαση σε υποδομές εύρος νομοθεσίας και κυρώσεις όλα αυτά συζητήθηκαν περαιτέρω πρόοδος επετέφθη ένας αριθμός πολιτικών θεμάτων πρέπει να επανεξεταστούν και να συζητηθούν περαιτέρω. Ο επόμενος τριμερής διάλογος θα διεξαχθεί αύριο και αναμένουμε λοιπόν αυτό να γίνει και για το, την, το τριμερή διάλογο που έγινε στο Στρασβούργο έγινε, σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την κατάρτιση και τα ερευνητικά ε, μέσα και σε σχέση με τον καθορισμό των ε, ε, αδικημάτων, κυρώσεις ε, και ποινές, δημοσίευση, δημοσιοποίηση αυτών των κυρώσεων και τα σχετικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο περαιτέρω τριμερή διάλογο που να προβλέπεται και το Συμβούλιο προβλέπεται να επανέλθει στο Ευρωκοινοβούλιο μετά την έκβαση της ομάδας εργασίας κατά την 16 Δεκεμβρίου και ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθούν οι εργασίες σε αυτό το σημείο χωρίς περαιτέρω τριμερείς διαλόγους. Αυτό είναι η ενημέρωση με τα στοιχεία από πλευράς ανακοινώσεων Προέδρου. Και μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες τώρα. Εσείς τι λέτε, παρακαλώ. Ε, ε Ωραία, Ελίζα, εσείς για τεχνικά προβλήματα ίσως τελευταία στιγμής θα μπορούσα να ζητήσω να αναβάλουμε για τρια 4 λεπτά την ψηφοφορία γιατί πρέπει κάποιες λεπτομέρειες να εξετάσουμε. Λοιπόν, κάποιες, ένα τελευταίο χτένισμα για, πριν από την τελική ψηφοφορία μπορεί να γίνει λοιπόν. Είσαστε έτοιμοι. Members put their για να κάνουμε μια δοκιμαστική πρώτα ψηφοφορία. Άρχεται η δοκιμαστική ψηφοφορία. Δοκιμάζουμε τις συσκευές και τις κάρτες. Άρχεται η ψηφοφορία για τη δοκιμαστική μας ψηφοφορία. 41, 41 μέλη παρόντα, 43 μέλη παρόντα, 38 έχουν πατήσει τα κουμπιά, 39, 40 τώρα. Τρία μέλη δεν πάτησαν τα κουμπιά των συσκευών τους, δύο δεν έχουν πατήσει τα κουμπιά των συσκευών τους. Πάντα με ανησυχεί βλέπετε αυτό όταν κάποιος δεν έχει, δεν έχει πατήσει το κουμπί της συσκευής του. Λοιπόν, όλοι τα πατήσατε, λειτουργούν οι συσκευές. Λοιπόν, πολύ ωραία. <clears throat> Οι 30 είναι ικανοποιημένοι, οι 8 όχι, οι 2 είναι αναποφάσιστοι, αποχές. Μάλιστα. are you asking for the floor? Ζητείτε να παρέμβετε εσείς. Πριν ξεκινήσουμε με το, AS, με το SRM να κάνω μια παρατήρηση αν μου επιτρέπετε για το SRM διότι κάποιες τελευταίες συζητήσεις που έγιναν με τις συναδέλφου για το εύρο, το φάσμα, αν μου επιτρέπατε θα ήθελα να διαβάσω, να σας αναγνώσω δύο προτάσεις για να υπάρξει μια διευκρίνηση. Διότι τι συμβαίνει με το SSM το SRM καλύπτει όλες τις τράπεζες επίσης, όμως στην πρακτική καθημερινή δουλειά οι εθνικές αρχές θα εκτελούν έργο όσον αφορά την σύνταξη ε, για προγράμματα και θέματα επίλυσης, ε, resolution κτλ. Όταν πρόκειται όμως για αποφάσεις ε, τέτοιου είδους και ιδιαίτερα όταν συμπεριλαμβάνεται η χρήση του Ταμείου, τότε αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται από το Συμβούλιο της ε, ενιαίας ε, εποπτικής αρχής και έτσι θα πρέπει αυτό να λαμβάνεται υπόψη επίσης. Okay, thank you Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν και μία ή δύο προφορικές τροποποιήσεις ε, και που θα πρέπει να τις διαβάσουμε όταν θα φτάσει η ώρα να ψηφιστούν. Ελπίζω ότι οι ομάδες θα είναι σε θέση να δώσουν, να έχουν αποσαφηνίσει αυτά τα πράγματα επαρκώς. Είσαστε έτοιμοι λοιπόν, ξεκινάμε. Τροπολογία 83 πρώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Συμβιβασμός α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός Β υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός Σ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός Δ, Πρώτα απ' όλα έχουμε μια προφορική τροποποίηση από την ECR να προσθεθεί η διατύπωση και η Επιτροπή. Όσοι είναι υπέρ αυτής της προφορικής τροποποίησης κατά αποχές απορρίφθηκε η προφορική τροποποίηση. Ο αρχικός συμβιβασμός D υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός τώρα ε, ή σε τμήματα ψηφοφορία, σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα, τι είπατε, θέλετε να ελέγξουμε το 2, το αποτέλεσμα για το, την ψήφιση του τμήματος 2. Συγγνώμη που πήγα πολύ γρήγορα. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε το 2. Ψηφίσατε όλοι. Εντάξει. 24 υπέρ 21 εναντίον εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 307. Μόλις την βρω. Εντάξει. 307 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός έφε Θα ελέγξουμε την 307 αν θέλετε. Αλλά ήταν σαφές νομίζω το αποτέλεσμα. Νομίζω το ΕΛΚ ήταν μόνοι τους ή του ΕΛΚ. Με άλλα λόγια. Ψηφίσατε όλοι. Δύο ακόμα πρέπει να ψηφίσουν. Λίγη τώρα η ψηφοφορία. Σε λίγο έληξε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 24 εναντίον 19 υπέρ. Συμβασμός F, σίγμα τάφ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβιβασμός G υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός G α υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 301, 381 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβασμός H υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός I υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. J Συμβιβασμό υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. K υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. L Συμβιβασμό L υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. M υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. N Πρώτα απ' όλα υπάρχει προφορική τροποποίηση του ΕΛΚ και των Πρασίνων. Είναι η προφορική τροποποίηση μόνο που ψηφίζουμε υπέρ, κατά, απόχες. Λοιπόν, να ελέγξουμε σε σχέση με την προφορική τροποποίηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίες. Η προφορική τροποποίηση εγκρίθηκε λοιπόν. Και τώρα θα ψηφίσουμε τον συμβιβασμό εν όπως τροποποιήθηκε από την προφορική τροποποίηση υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε νομίζω με την ίδια πλειοψηφία και περνάμε τώρα στον συμβιβασμό ο όμικρον. Σε τμήματα ψηφοφορία. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε το δεύτερο. Περνάμε τώρα στην 587 τροπολογία. Πώς είπατε εσείς? Εντάξει. 587 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβασμός π υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Q υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε R Α, είναι νέα σε τμήματα ψηφοφορία. Λοιπόν, προετοιμαστείτε, θα σας διαβάσω περί πρόκειται. Το έχω σε δύο τμήματα εγώ. Πρώτο τμήμα. Όσοι είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε περνάμε στο συμβιβασμό S υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε T υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε U υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 643 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Β υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 649 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έχουμε σε τμήματα ψηφοφορία στη συνέχεια α έχουμε τώρα έχουν, έχει αποσυρθεί δεν θα ψηφιστεί αυτό ο συμβασμός W τώρα ωραία ωραία αποσύρθηκε για τον συμβιβασμό είχε υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται συμβιβασμός 6 που βρίσκεται σελίδα 35 συμβιβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Y υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Y α υπέρ μια στιγμή δημιουργήθηκε κάποια σύγχυση Πολ είσαι εναντίον υπέρ Λοιπόν, θα το κάνουμε ηλεκτρονικά, ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. YA, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. YA. YA. Δεν φοράω τα γυαλιά μου σήμερα και είναι δύσκολο να διακρίνω ακριβώς τι γίνεται κάτω στην αίθουσα. Λοιπόν, ωραία, απορρίφθηκε το YA, YA. Ωραία. Δεν νομίζω με μία ψήφο διαφορά να είχαμε άλλο αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάει, απορρίφθηκε. Συμβιβασμό Z υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στο ΑΑ συμβιβασμό υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμό ΑΒ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 731 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίφθηκε. AC συμβιβασμός υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 732 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Συγγνώμη Παύλο, ήταν και δική σου αυτή, μάλιστα. AD συμβιβασμός με προφορική τροποποίηση ECR. Έχετε, θα πάρουμε πρώτα αυτή την προφορική τροποποίηση. Όσοι είναι υπέρ αυτής, κατά αποχές. Η προφορική τροποποίηση απορρίφθηκε. Έτσι λοιπόν ο συμβιβασμός AD ως είχε αρχικά υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβιβασμός AE, αε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. AF, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. AG, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. AH υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε AI υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε AJ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε AK υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε AL υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε AM υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε AN υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε AO υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε AP υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε AQ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε AR υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε AS υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε AT υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. AU υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. AV υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. AW σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. AX υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε AY υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 877 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβασμός BA υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε BB υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Τοπολογία 882 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. BC ε, συμβιβαστική τροπολογία. BC υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. BD υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. BE υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. BF υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε BG υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε BH υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε BI έχουμε μια προφορική τροποποίηση της ECR πρώτα αυτή υπέρ της προφορικής τροποποίησης κατά αποχές απορρίφθηκε η προφορική τροποποίηση πάμε στο συμβασμό BI όπως είχε αρχικά υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε BJ συμβασμός υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε BK υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε BL υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε BM υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε BN υπέρ BN υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε BO υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε BP σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε το δεύτερο τμήμα πάμε τώρα στο συμβασμό BQ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε BQ α υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. BS υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τώρα τροπολογία 1019 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. BT συμβιβασμός υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. BU υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. BV υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. BW υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε BX υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε BY υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε BZ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός CA υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε εντάξει τώρα. Αύκο 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 87 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. CB συμβασμός υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. CC υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η CC τροπολογία 90. Πώς είπατε? Α, συγγνώμη, εντάξει, μάλιστα. Πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 89 τώρα, υπέρ. Πρώτα η 89. Ναι, γιατί ο συμβιβασμό CC καταψηφίστηκε. Ψηφίζουμε την τροπολογία 89, υπέρ. Κατά. Δεν θα ελέγξουμε γιατί δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Εντάξει, ψηφίζουμε την 89. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι στο γκρι χρώμα συμβιβασμός επειδή καταψηφίστηκε ο συμβασμός CC. Τροπολογία 89. 5, 4, 3, 1 να ψηφίσει. Κλείνει η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Απορρίφθηκε η 89. Πάμε στην τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτή απορρίφθηκε. Και τώρα η τροπολογία 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 90 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Λοιπόν, ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Πράγματι είχε εγκριθεί. Εγκρίθηκε λοιπόν η 90. 91 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. CD συμβιβασμός υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. CE υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. CF υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. CG υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. CH υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 98 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 97 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Συμβασμό CHα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε CI υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε CJ σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 103 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 104 υπέρ κατά α, θα ελέγξουμε την 104. Ψηφίζουμε την 104 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας και απορρίφθηκε. Η 105 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε CK υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε CR υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε CM υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε CN υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε CO υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε 123 τροπολογία υπέρ κατά άποχες απορρίφθηκε Εντάξει, θα ελέγξουμε για την 123, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εντάξει, πολύ καλά. Λοιπόν, όχι, η 123, τέλος ψηφοφορίας τώρα. Νομίζω σωστά το είχαμε πει ότι καταψηφίστηκε. Πέρα ψηφοφορία, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα, είχε απορριφθεί, απορρίφθηκε. Πάει. Μικρή διαφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Το κάναμε μόλις Εντάξει, πολύ καλά. Πολλές, πολύ πανηγυρίσαμε λοιπόν μετά από αυτό. Τέλος πάντων, ωραία. Τροπολογία CP υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. CQ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. CQα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. CR υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε αύκο 5 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε την αύκο 5 ψηφίζοντας ηλεκτρονικά νομίζω εγκρίθηκε αλλά έρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας και πράγματι εγκρίθηκε λοιπόν CS τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. CT υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. CV υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. CW υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. CWα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. ΑΦΚΟ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. CX υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. CY υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. CZ υπέρ κατά αποχές. Θα ελέγξουμε την CZ. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Δεν έχει λήξει η ψηφοφορία ακόμα, μια στιγμή. Ή απορρίφθηκε, μάλιστα, πολύ καλά δεν υπάρχει κάποιο θέμα να ψήφισε κάποιος λάθος ή να έγινε λάθος, απορρίφθηκε, τελείω και παύλα. Πάμε τώρα και ψηφίζουμε την 158 τροπολογία υπέρ. 158 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίφθηκε αυτή. Η 146 υπέρ. Κατά. Απόχες. Και αυτή απορρίφθηκε. Πάμε στο συμβιβασμό DA υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Αύκο 9 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την ΑΦΚΟ 9. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Και πράγματι απορρίφθηκε. Πάμε στην τροπολογία DB. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 10 άρχεται η ψηφοφορία ένας ακόμα να ψηφίσει τώρα θα κλείσει η ψηφοφορία έκλεισε η ψηφοφορία αποτέλεσμα απορρίφθηκε η 156 και η 11 αύκο υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκαν. DC τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. DD υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. DE υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 162 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 163 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. DF υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε DG υπέρ κατά απόχες να ελέγξουμε ψηφίζουμε την DG ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία Τώρα θα λήξει η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Λοιπόν, εγκρίθηκε με μία ψηφοδιαφορά Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στην DH υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε DI υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε DJ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε DK υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε DL υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε DM υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε DN υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε DO υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε DP υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε DQ Πρώτα απ' όλα προφορική τροποποίηση της CCR Υπέρ της προφορικής τροποποίησης, παρακαλώ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την προφορική τροποποίηση ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ένας να ψηφίσει ακόμα για να ολοκληρώσουμε. Κλείνει η ψηφοφορία. Λοιπόν, καταψηφίστηκε. DQ τώρα, στο αρχικό κείμενο. DQ, χωρίς τροποποίηση, υπέρ. Κατά, απόχες, εγκρίθηκε. DR υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε DS υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε DT υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε DT α υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε DU υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε DV υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε DV α υπέρ Μάλιστα. DV α υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. DW υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. DX υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 197 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. DY υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. DZ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 200 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 201 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία EA υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε πάμε τώρα στις τροπολογίες που ακολουθούν οι 16 και οι 202 υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν. EB τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. EC υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. ED υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. ED α υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Μάλιστα ωραία να ελέγξουμε. EDA ελέγχουμε. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε άρχεται. Συγγνώμη προφανώς ε, δεν το αντελήθη σωστά. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορία. Ωραία και πράγματι απορρίφθηκε. Ωραία. Πάμε λοιπόν στην τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτή απορρίφθηκε. Η 207 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτή απορρίφθηκε. Πάμε στην ΙΙ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η F σε τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 212 όχι λάθος EG τροπολογία EG υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 212 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 213 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε και αυτή EH υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε EI υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε EJ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε EK υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η L υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η ΕΜ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Λοιπόν, τώρα ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Δύο ακόμα για να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, λίγη τώρα η ψηφοφορία. Κάποιος δεν πάτησε το κουμπί του, εντάξει, λίγη η ψηφοφορία. 34 υπέρ, 3 εναντίον, 8 αποχές. Και ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Ψηφίσατε όλοι. Τρει ακόμη. Λίγη σε λίγο η ψηφοφορία. Λίγη. Έληξε. Λοιπόν, 35 υπέρ. 2 εναντίον. Και 7 αποχές. Πολύ καλά. Λοιπόν, εισηγητά, θέλετε να παρέμβετε. Να, να ψηφίσουμε την απόφαση για να ολοκληρωθούν να ε, διαπραγματεύσουμε το Συμβούλιο, να τερματιστούν. Λοιπόν, απόφαση για τις διαπραγματεύσεις για την πρώτη ανάγνωση με την κανονική σύνθεση. Πρέπει να ψηφίσουμε επ' αυτού για να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Άρχεται. Ένας ακόμα να ψηφίσει. Ψηφίζουμε ακόμα. Λίγη ψηφοφορία σε λίγο. Λοιπόν, έληξε 38 υπέρ, 5 εναντίον, 2 αποχές. Λοιπόν, θα αρχίσουμε διαπραγματεύσεις με την ομάδα μας, με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ, συγχαρητήρια σε όλους σας. I, Ελίζα, δεν θέλω να καθυστερήσουμε περισσότερο με την ψηφοφορία, αλλά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο συμβαστικό πνεύμα, όχι μόνο των εισηγητών, αλλά όλων των μελών, όλων των αντιπροσωπιών, γιατί έτσι έχουμε μια ισχυρή θέση απέναντι στο Συμβούλιο για τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η ψηφοφορία αυτή ήταν πολύ σημαντική και ελπίζω και εγώ το Συμβούλιο να λάβει υπόψη του τη γραμμή που υιοθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να καταλάβει ότι δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ για κυβερνητική μέθοδος όπως αυτούς. Προχωράμε. Ερχόμαστε στο Ζων Πολ Τροπολογία αριθμό 2. Τροπολογία αριθμός 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία αριθμός 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη φοφορίες. «42 υπέρ, καμία ψήφος κατά και δύο αποχές». Ψηφίζουμε τώρα το νομοθετικό κείμενο. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της φοφορίες. 42 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά και δύο αποχές. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε και περνάμε τώρα στο σημείο 14. Για το σημείο 14 δεν έχω κατάλογο, λέει η Πρόεδρος. Σέμπο Τέρο. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική γάμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική δέλτα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, υπέρ 29, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική F σιγματάφ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. G σε δύο τμήματα. Ζ, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με δύο ψήφους διαφορά, συγγνώμη. 37 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ για την 37. Ψηφίσατε όλοι. πέρα της φοφορίας. Απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική ήττα. Υπέρ. Κατά. Α, είναι κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική I, θ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική J, ι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται και η υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. «57 υπέρ». Α, μια στιγμή. Μπερδεύομαι με τις σελίδες. Όταν λέω σελίδα μπερδεύομαι. Λοιπόν, 58 υπέρ, κατά, Ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 58. Ψηφίσατε όλοι. Όχι, εγώ δεν ψήφισα. Ήμουν αφηρημένη, λέει η πρόεδρος. 58 ήταν, έτσι, ναι. 61 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 62. Καλά. Συγγνώμη. 61. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεν κοίταζα καλά μάλλον. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 21 ψήφι υπέρ, 24 κατά. 62 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε για την 62 νομίζω την κρίνεται αλλά για να δούμε ψηφίστε παρακαλώ ψηφίσατε όλοι πέρα στις φοφορίες εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Αν δεν με πιστεύετε, να ελέγξουμε. Απορρίφθηκε, πράγματι. 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο, 16 παράγραφος υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψη α υπέρ. Δεν υπάρχουν τροπολογίες, είναι το αρχικό κείμενο της αιτιολογικής σκέψης α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπάρχει προφορική τροποποίηση του συγκητή να αλλάξει μια φράση. Πρώτα την προφορική τροποποίηση ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Συνεπώς τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία, την αρχική τροπολογία, αριθμός 1. Τι θέλετε, να ελέγξουμε για την προφορική τροποποίηση. Ωραία. Δεν βλέπω τι ότι 22 «22-22». Απορρίπτεται. Δεν ήταν σαφέ, πράγματι. Τώρα λοιπόν ψηφίζουμε χωρί την προφορική τροποποίηση τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τώρα τροπολογία 2 υπέρ, υπέρ, τροπολογία 2, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, να κρατάτε τα χέρια σας ψηλά. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται νομίζω. Καλά, θα ελέγξουμε αν θέλετε. απορρίφθηκε. Κάποιοι εξαφανίζονται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά ηλεκτρονικά θα ελέγξουμε για την 9 γιατί κάποιους εδώ σας χάνω εγώ τουλάχιστον τα έχω χάσει μάλλον λέει η πρόεδρος λοιπόν κοντεύουμε κοντεύουμε πέρα της φοφορίας Α, καλά. Εντάξει, δεν είναι απλώς κάποιες αμφιβολίες, τέλος πάντων. Όντως. Ε, τώρα, τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο της σιγματάφ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 12 είναι συμβατή υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το τροποποιημένο κείμενο ηλεκτρονικά παρακαλώ. Κοντεύουμε να τελειώσουμε. Το αποτέλεσμα 44 υπέρ, καμία ψήφος κατά και δύο αποχές. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο κύριε Τεύκο. Τώρα ψηφίζουμε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ε? Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ, κατά αποχ... Δεν είμαι σίγουρη. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 3 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είδα κανέναν από το ΕΛΚ να σηκώνει το χέρι του. Μάλιστα. Ωραία, εγκρίνεται, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 6, άρτη ψηφοφορία. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Τρεις ακόμη πρέπει να ψηφίσουν. Πέρας. Απορρίπτεται σαφώς. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Συγγνώμη. Και για την προηγούμενη τροπολογία ήταν αυτό. Είμαστε πλέον τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση και το πρώτο τμήμα της 8 νομίζω ότι εγκρίνεται, λέει ο Πρόεδρος. Ψηφίσατε όλοι πέρας, όντως εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 8 υπέρ,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 Όντως εγκρίνεται. Περνάμε στην παράγραφο 9, τροπολογία 17, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά αποχές Σηκώστε χέρια σας παρακαλώ πολύ για την 18, ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία υπαριθμών 18. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 20 παρακαλώ πέρας Πέρας της πληροφορίας. Και εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τροποποιημένο κείμενο. άρθρο ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Πρωτού φύγετε όλοι. 39 υπέρ μία ψήφος κατά και μία αποχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε τίποτα άλλο στην ημερήσια διάταξη. Η επόμενη συνεδρία είναι σε 9 Ιανουαρίου, σε 9 η ώρα το πρωί. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ.